συνεδρίαση της 17ης ε, Δεκεμβρίου και με λύπη σας ε, πληροφορώ πως η Πίλαρ Χουάρες Μποά, η υποδιευθύντρια της ε, αποστολής μας στην ΑΕΤ, εξακολουθεί να αγνοείται. αναζητείτε ακόμα η Πίλαρ ήταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως ε, σήμερα η σκέψη μας πηγαίνει στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτή την ε, τραγωδία. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναγγείλει πώς θα στείλουν σημαντική οικονομική βοήθεια και 150 αστυνομικούς μεταξύ άλλων. Πολλά κράτη-μέλη έστειλαν και ε, άλλη βοήθεια. Είναι, μια, είναι η σημαντικότερη καταστροφή στην ιστορία της Αιτής και μία από τις ε, σημαντικότερες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αγνοούνται επίσης πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Z Επίσης ε, με λύπη πληροφορήθηκα την εκτέλεση του Εγνάς Σακύρ ε, Βρετανού υπήκου ο οποίος εκτελέστηκε στην Κίνα ε, εκτελούνται γύρω στα 7.000 άτομα στην Κίνα κάθε έτος πρόκειται για τον πρώτο Ευρωπαίο πολίτη από το 1951 που εκτελέστηκε στην Κίνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει όπως πάντα την επιβολή της ανατικής ε, ποινής ε, και θέλουμε να γίνει μια πιο λεπτομερής έρευνα για την εκτέλεση αυτή. Χθε επίση. είχαμε τον πρώτο γύρο πολιτικών εκλογών στην ε, Ουκρανία. Συνάδελφοί μας ήταν παρατηρητές επιτόπου. Δεν έχουμε ακόμα επίσημες πληροφορίε όσον αφορά την διεξαγωγή των εκλογών. Οι συνάδελφοι δεν